I Ας προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε με τις επεξηγήσεις ψήφου. Πρώτον, επί της εκθέσεως Μπέγκε, έχω την κυρία Οβέ ως πρώτο όνομα. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λίγο δύσκολο να μιλήσω με αυτό το θόρυβο, αλλά η υλοποίηση ε, του μηχανισμού αυτού και η απόφαση που λάβαμε δείχνει πόσο επιτυχής ήταν η συνεργασία των θεσμικών οργάνων. Δείχνει επίσης ότι κρίνουν τα θεσμικά όργανα ότι είναι απαραίτητη χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος. Κάτι άλλο σημαντικό ήταν ότι πετύχαμε να βρούμε τον κρίκο της αλυσίδας που έλειπε σε τα ενεργειακά προγράμματα. Uh, Επόμενη έκθεση, επίσης του κυρίου Μπέγκε για το σχέδιο για την ανάκαψη της οικονομίας σε ίδια ομιλήτρια. Ε, τένον, συγκασέτα ράπορτιτ. Κυρία Πρόεδρε, υποστήριξα και αυτή την ε, έκθεση το αποτέλεσμα της Επιτροπής Συνδιαλλαγής, κατά την άποψή μου, ήταν θετικό. Ξέρετε ότι η διαδικασία ήταν περίπλοκη, αλλά το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικά θετικό. Υιοθετήθηκε το πρόγραμμα ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για τον προϋπολογισμό, δώσαμε 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ για το στόχο αυτό. Υποστήριξα λοιπόν και αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Εκθέση Σιριάν Μάνκα. Ο κύριος Ντέιβις πρώτος μιλήτης, για την επεξήγηση ψήφου. Ο κύριος Γκρίφιν από το British National Party ε, άφησε να υπονοηθεί ότι ψήφισε λόγω, όπως ψήφισε λόγω ε, προσωπικών ε, συμφερόντων. Εγώ ουδέποτε έκανα, έλαβα χρήματα για τη δουλειά που κάνω καταπολεμώντας τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Όλα τα έσοδα που έλαβα περιλαμβάνονταν στις δηλώσεις συμφερόντων. Αυτό δεν με εμποδίσει ωστόσο ποτέ να καταγγέλω κάποια προγράμματα που είναι τελείως αερολογίες. Καθ' όλη τη διάρκεια της μου ο κύριος, ε, αγωνιζόμουν με βάση τις αρχές μου, ο κύριος Γκρίφιν ας εξηγήσει γιατί το κόμμα που, το οποίο ηγείται ο ίδιος δύο φορές δεν υπέβαλε εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς στην, στην, Ευρω... Βρετανική Εκλογική Επιτροπή που ούτως ή άλλως δεν δείχνουν σωστά την, κατάσταση, την οικονομική κατάσταση του κόμματός του. Πολλοί υποψιάζονται ότι πολλά μέλη του κόμματός του χρησιμοποίησαν την, ε, τα κονδύλια του κόμματος για προσωπικούς στόχους. Ας δώσει λοιπόν κάποιους, ε, κάποιους ε, ο, λογαριασμούς ο κύριος Γκρίφιν που θα εγκρίνουν οι λογιστές. Ο κύριος Φόξ κατόπιν. Πρόεδρε, να πω ότι ο Τζόιν Ντόνιγκ, ένας ε, Βρετανό ε, βουλευτής ε, του 18ου αιώνα, είπε και παραφράζω ότι αυξάνεται ο προπολογισμό και θα συνεχίσει να αυξάνεται. Δεν πρέπει να μειωθεί. Εγώ καταψήφισα γιατί υπερβαίνει το όριο του 1% για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Αυτό το όριο δεν θα πρέπει να υπερβληθεί. Θα πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι κάθε ευρώ το οποίο ξοδεύουμε είναι ευρώ του φορολογούμενου και θα πρέπει να είμαστε συνετοί με τα χρήματα αυτά και ο προπολογισμό αυτό δεν ήταν συνετό. Ο κ. Καμάου, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και είναι υπέροχο να τελειώνουμε στα στιβαρά σας χέρια το χρόνο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πάρω το λόγο και να σας ξαναδώ. Θα ήθελα να πω ότι και εγώ, όπω ο προηγούμενο συνάδελφο, καταψήφισα τον προπολογισμό. Πολύ συχνά μιλάμε για κοινέ ευρωπαϊκέ αξίε και αλληλεγγύη. Ωστόσο, σε μία στιγμή που πολλέ κοινότητε, πολλέ οικογένειε πλήττονται από την οικονομική κρίση, αγωνίζονται να πληρώσουν του λογαριασμού, χάνουν τι δουλειέ του, περικόπτονται οι μισθοί, είναι νομίζω έξωφρενικό να ψηφίζουμε για να αυξηθεί ο προπολογισμό που δεν λαμβάνει υπόψη καθόλου την τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Χρειαζόμαστε σωστά δημοσιονομικά. Θα πρέπει να κατανοήσουμε και να το δείξουμε ότι κατανοούμε τις ανησυχίες των, ε, του εκλογικού μας σώματος. Μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε την ανάπτυξη η οποία χρειάζεται ε, για να βοηθήσουμε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό καταψήφισα τον προϋπολογισμό και θα ήθελα να σας ευχηθώ ε, καλά Χριστούγεννα και τυχισμένο το καινούργιο έτος. Ευχαριστώ και τώρα να περάσουμε στην έκθεση για τη Λευκορωσία, λέει η Πρόεδρος, η κυρία Αντρικάιναν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του ψηφίσματος, γιατί η Λευκορωσία σήμερα καταδεικνύει ένα επίπεδο δέσμευση σε ό,τι αφορά την συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά από τις πολλέ συζητήσει ε, με την Λευκορωσία είναι περιορισμένα τα αποτελέσματα. Πρόσφατα ακούσαμε από την αντιπολιτευσή ότι ο πρόεδρος σκοπεύει να υπογράψει ένα διάταγμα που θα ε, περιλαμβάνει την ε, θα περιορίζει την πρόσβαση στο διαδικτύο και στην ελεύθερη ενημέρωση. Θα πρέπει να προσελκύσουμε την ε, Λευκορωσία πιο κοντά στην Ένωση. Αλλά καταρχάς θα πρέπει να προσεγγίσουμε τον λαό της Λευκορωσίας γιατί τώρα φαίνεται ότι μιλάμε με τις αρχές της Λευκορωσίας. Ε, αυτό που χρειαζόμαστε είναι προσέγγιση ε, της Λευκορωσίας. Είναι πολύ ακριβή η θεώρηση σε ύψους 60 ευρώ για να έρθει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. δεν θα ε, επλήττονταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αν η βίζα αυτή κάλεπτε μόνο τα έξοδα, τα 5 ευρώ δηλαδή, για την θεώρηση. Θα ήθελα να παρακαλέσω, λέει η Πρόεδρο, τον κύριο Σάρο και τον κύριο Μπρόκ να βγουν έξω να συνεχίσουν τι συζητήσει του. Μα κύριε Μπρόκ, έξω, έξω σας παρακαλώ τους καυγάδε σα. Could you please have your... Σας παρακαλώ, τις συζητήσεις σας έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας. Out. Mr. Brock, will you please... Μα κύριε Μπροκ, μπορείτε να βγείτε έξω, να συνεχίσετε τη συζήτησή σας. Κύριε Πρέντα, αν θέλετε να κάνετε επεξήγηση ψήφου, θα σας ακούσω τώρα για τη Λευκορωσία. Αυτό επιθυμείτε? Ευχαριστώ. Να ζητήσω επεξήγηση ψήφου για την πρώτη πρόταση του κυρίου Σούλτς. Δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτή η πρόταση. Θα ήθελα απλά να εξηγήσω γιατί ψήφισα έτσι για την πρώτη πρόταση του κ. Σούλτ. Λυπάμαι, δεν είναι δυνατόν. Νόμιζα ότι θέλατε να μιλήσετε για την έκθεση για τη Λευκορωσία. Και τώρα περνάμε στον κατάλογο για το ψήφισμα για την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η κυρία Αντρεκάνιον και πάλι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματο, γιατί η κατάσταση στο Κονγκό είναι φρικτή. Δεκάδες χιλιάδες ε, θάνατοι ε, στην επαρχία κάθε μήνα λόγω της βίας από τις ε, στρατιωτικές ομάδες. Χρησιμοποιείται αδιακρίτως η βία και πολλές φορές θύματα της πέφτουν και άμαχοι πολίτες απλοί. Πραγματικά και η κατάσταση κατά των γυναικών, ε, η σεξουαλική βία ε, είναι αποτρόπαιη. Και όλοι οι πλευρές είναι υπεύθυνες για αυτή την κατάσταση και ο στρατός. Η αστυνομική αποστολή είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί το βασικό πρόβλημα που υπάρχει είναι τα φαινόμενα ατιμορρησίας ε, στο Κονγκό και οι συνεχείς πράξεις καταστολής ε, και βίας. Όπως και στη Ρουάντα μπορεί η αστυνομική δύναμη να επιτύχει ε, στην περιοχή αυτή. Πρέπει λοιπόν με περισσότερη δράση να γίνει, πρέπει να δοθούν και περισσότεροι πόροι μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ. Και τέλος ο κύριος Ντέβα a few minutes ago. Madam Όπως ε, όσο πλέον πλησιάζουν οι χριστιανικές διακοπές, ε, μας περιμένουν οι παχές γαλοπούλες, τέλο πάντων ό,τι άλλο τρώει ο καθής ε, από εμάς ενορταστική περίοδο, ε, ακούμε ότι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό πολλά άτομα θα πεθάνουν την περίοδο αυτή ακριβώς που εμείς θα γιορτάζουμε. Σχεδόν 5 εκατομμύρια έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους μετά, από το 99 και μετά στη χώρα αυτή. Και εκτιμάται ότι 45.000, όσο δηλαδή μια μικρή βρετανική κομμόπολη, πόλη, 45.000 άτομα ε, χάνουν τη ζωή τους, σκοτώνονται κάθε μήνα. Γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Δεν θα έπρεπε να σκεφτόμαστε το, τη μοίρα αυτού του λαού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Γιατί ξέρετε, στον ίδιο πλανήτη ζούμε όλοι μας. Για πάνω από 20 χρόνια τα Ηνωμένα Έθνη με σθένος και κουράγιο προσπαθούν ε, να σταθεροποιήσουν κάπως την κατάσταση. Όμως έχουν μόνο 20.000 στρατιώτες επί τόπου. Πώς μπορεί να διατηρηθεί η ειρήνη με 20.000 στρατιώτες μόνο. Πρέπει να βοηθήσουμε τον ΟΗΕ να κάνει αποτελεσματικά τη δουλειά του και τα άτομα τα οποία δρούν ατιμόρυτα, που βιάζουν και σκοτώνουν γυναίκες και παιδιά, πρέπει να σταματήσουν. Κάποιος να τα σταματήσει αυτά τα φαινόμενα και αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Ευχαριστώ. Η πρόεδρος, αυτό ήταν, αυτός ήταν ο τελευταίος ομιλητή στον κατάλογο μιλητών. Εάν κάποιος θέλει να κάνει επεξήγηση ψήφου, ε, πρέπει, όπως γνωρίζετε, να έχει ενημερώσει και τον προτέρων τη γραμματεία. Σας βλέπω, ε, κύριε Μπουζούτιλ, κάτι σας ανησυχεί. Κυρία Πρόεδρε, ζήτησα επεξήγηση ψήφου για το ψήφισμα για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για την πρόσβαση στα έγγραφα μετά τη θέση και τη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά μάλλον δεν ε, λάβατε το αίτημά μου. Πρόεδρος, μάλλον υπήρξε κάποιο ασύνηθες ε, σφάλμα στην όλη διαδικασία και πράγματι δεν λάβαμε το αίτημα. Μπορείτε λοιπόν να προχωρήσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους του ΕΛΚ θα ήθελα να τονίσω ότι το ΕΛΚ καταψήφισε το ψήφισμα όχι γιατί δεν είναι υπέρ της διαφάνειας ή της πρόσβασης στα έγγραφα. Φυσικά ε, το αντίθετο ισχύει στο πλαίσιο της ε, νέας συνθήκης που τέθηκε σε ισχύ. Απλά ε, ψηφίσαμε, θα θέλαμε να είχαμε ψηφίσει το δικό μας ψήφισμα σε αυτού, πέρα αυτού του ψηφίσματος ήμασταν, διότι θεωρούμε ότι ε, ακολουθεί μια πιο σωροπημένη προσέγγιση για το λεπτό αυτό ζήτημα. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν συζητούμε το ζήτημα τη διαφάνεια και τη πρόσβαση στα έγγραφα ώστε να μην ξεπεράσουμε κάποια όρια και να μην εκθέτουμε έγγραφα και διαδικασίες σε βαθμό που καθιστά μη δυνατόν να λειτουργήσει το όλο σύστημα. Γιατί κάποιες φορές μπορούμε κλείνοντας τις διαπραγματεύσεις, ε, μάλλον αποκαλύπτοντας τα πάντα για κάποιες διαπραγματεύσεις, τελικά να τις ε, παρακολύσουμε και να τις καταστρέψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λέει Πρόεδρος, εδώ ολοκληρώνονται οι εργασίε ε, για την πρωινή σύνοδο και θα επανέλθουμε στις 3 το μεσημέρι.